Είναι μια πρωτοβουλία της Επιτροπής Απασχόλησης Ελληνικών Υποθέσεων. Δίνω το λόγο στην κυρία Ουρσκοκ που συνέταξε το κείμενο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κρίση έχει προκαλέσει την άνοδο της απασχόλησης των νέων σε σχετικά επίπεδα. Πολλοί νέοι δεν έχουν ε, και δεν καταφέρνουν να βρουν την πρώτη τους δουλειά και έτσι να πετύχουν ανεξαρτησία στη ζωή τους. Το 2013 για να βοηθηθεί και να ε, απαρενθεί το πρόβλημα αυτό, δημιουργήθηκε η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, για να δοθεί απασχόληση και να προωθηθεί η απασχόληση των νέων στις πιο πληττόμενες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ άλλων με προγράμματα εγγύησεων για τους νέους. Και η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων ε, χρηματοδοτήθηκε από 1η Σεπτεμβρίου 2013. Αλλά μετά από ένα χρόνο και παραπάνω από την εφαρμογή του προγράμματος δεν ε, ανταποκρίνονται τα αποτελέσματα στις προσδοκίες. Η απορρόφηση των πόρων από τα κράτη-μέλη δεν έχουν οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση των ευκαιριών για την επασχόληση των το πρόβλημα. Η πρωτοβουλία προτάθηκε αρχικά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ωστόσο στην παρούσα φάση 1,5 χρόνο μετά από την χορήγηση των κονδυλίων, τα κράτη-μέλη και η χρήση των ε, κονδυλίων αυτή αυτών δεν ε, έχει επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα πέρα από την έλλειψη χρηματοδότησης και ρευστότητα για την πρωτοβουλία απασχόλησης των νέων. Ετίθεται και ένα θέμα προχρηματοδότησης. Τι είναι αυτό που εμποδίζει τα κράτη-μέλη και τι σκοπεύει να κάνει το Συμβούλιο προκειμένου να πετύχει την επιτυχή και γρήγορη εφαρμογή. Τα κράτη-μέλη που έχουν την μεγαλύτερη, τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας των νέων και τα οποία έχουν πληχθεί πιο πολύ από την κρίση είναι αυτά που αντιμετωπίζουν και τα μεγαλύτερα προβλήματα στην εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων για την απασχόληση των νέων. Ενώ ουσιαστικά χρειάζονται μακροπρόθεσμες πολιτικές. Τι προσκόμματα λοιπόν αντιμετωπίζουν και τι βελτιώσεις μπορεί να μας υποσχεθεί το Συμβούλιο. Μπορεί να μας ε, εγγυηθεί κάποια χρηματοδότηση το Συμβούλιο όταν, έχει, όταν τελειώσουν και τα κονδύλια front-loading. Το Κοινοβούλιο θέλει να χρησιμοποιηθεί σωστά και ποδοτικά τα κονδύλια προχρηματοδότησης προτού τεθεί σε εφαρμογή ως ειδικό κανονισμό. Τι μέτρα λοιπόν ε, οραματίζεται το Συμβούλιο προκειμένου να καθησυχάσει και το Κοινοβούλιο αλλά και τους νέους ανέργους. Πώς ε, σκοπεύει να απαλύνει τα προβλήματα των ε, νέων ανέργων. Το Συμβούλιο μπορεί να, υπογρα... μπορεί να υποσχεθεί μια αξιολόγηση της πρόοδου έξι μήνες μετά από την θέση σε εφαρμογή του τροποποιητικού διορθωτικού κανονισμού και πώς ε, θα αντιδράσει το Συμβούλιο αν τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά ακόμα και μετά από την αύξηση της προχρηματοδότησης. Ευχαριστούμε και τώρα το λόγο έχει η κυρία Καλίνια Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Χαίρομαι για την ευκαιρία που μου δίνετε να συζητήσω μαζί σας την κατάσταση στην αγορά εργασίας για τους νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Προεδρία προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στη βελτίωση των συνθηκών υπό τις οποίες ε, μια μεγάλη κοινωνική ομάδα που είναι οι νέοι ε, έχουν πρόσβαση στην αγορά απασχόλησης. Αναφερόμαστε στους νέους και κυρίως στους νέους χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση και τα επαρκή προσόντα. Πρέπει να έχουμε ολοκλήρωση της αγοράς εργασίας. Αυτό παραμένει προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Στρατηγική Ευρώπη για το 2020 δίνει ιδιαίτερη σημασία στην υλοποίηση αποτελεσματικών μέτρων για την απασχόληση των νέων. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι η ανεργία των νέων παραμένει σε πολύ ψηλό επίπεδο, σε πολλά κράτη-μέλη. Έχουμε απώλεια ανθρωπίνων πόρων ουσιαστικά και καταστροφικές συνέπειες για το υπόλοιπο του εργασιακού βίου με την ανεργία των, θέων, των νέων. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν η πρωτοβουλία για την εγγύηση για τους νέους είναι εξαιρετικά σημαντική. Καταπολεμούμε την ανεργία των νέων στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο εκεί όπου η ανεργία των νέων είναι στο 25%. Ως ε, θετικό παράδειγμα, θέλω να υπογραμμίσω το, την εμπειρία της ε, Λετωνίας, η οποία ξεκίνησε να υλοποιεί την εγγύηση για τους νέους τον Ιανουάριο του 2014 και ήδη βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Η ανεργία των νέων έχει μειωθεί κατά 3,8% το 2014, μέσα σε ένα χρόνο. Πολλά εξαρτώνται από τα προγράμματα που εφαρμόζουν και υλοποιούν τα κράτη-μέλη. Παρ' όλα αυτά, είναι σαφές ότι παραπάνω πράγματα πρέπει να γίνουν. Παρά το ότι είναι μια ε, πολλά υποσχόμενη ενθάρρυνση, η πρωτοβουλία για τους νέους και η εγγύηση για τους νέους δεν μπορούν να λύσουν όλα τα προβλήματα. Είναι μέρος των εργαλείων, των, όλων των εργαλείων που υπάρχουν για να ε, λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Η χύτερη περίοδος εφαρμογής την της πρωτοβουλίας για την ανεργία των νέων σε σύγκριση με, τον, με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τους ε, ε οικονομικούς κύκλους σημαίνει ότι η πρώτη περίοδος θα είναι κρίσιμη για την επιτυχία του προγράμματος. Ε, εκατομμύρια Ευρωπαίοι ε, πρέπει να βρουν μια θέση απασχόλησης και δεν έχουν αρκετή πρόσβαση σε εκπαίδευση ή σε κατάρτιση. Είμαι πεπισμένη ότι τα αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμφωνούν με την άποψή μου. Ότι δηλαδή δεν πρέπει να καθυστερούμε άλλο, πρέπει να εφαρμόσουμε αμέσω την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Ιδαλλιώ θα πληγούν οι δράσει που έχουν ήδη αναλάβει τα κράτη-μέλη για να καταπολεμήσουν την ανεργία των νέων. Ένα από τα κύρια ε, εμπόδια είναι η έλλειψη επαρκών ταμιακών ροών για να, γίνουν, να καταβληθούν οι προκαταβολές στους δικαιούχους. Η Προεδρία θέλει να επιταχύνει το χρονοδιάγραμμα ε, για την προώθηση της νομοθετικής ε, πρότασης έτσι ώστε γρήγορα να εφαρμοστεί το να δίδεται χρηματοδότηση στα κράτη-μέλη σε πιο αρχικό στάδιο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ε, είναι προϋπόθεση για να έχουμε αυτά αποτελέσματα και μάλιστα γρήγορα. Συμφωνώ με όσους ε, υιοθετούν αυτή την άποψη. Αν έχουμε παρκή ρευστότητα κατά την αρχή της διαδικασίας υλοποίηση, τότε μπορούμε να υιοθετήσουμε τα πιο σχετικά μέτρα, της πολιτικής που μας ενδιαφέρουν περισσότερο. Μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι διότι η νομοθετική πρόταση που τροποποιεί την υφιστάμενη νομοθεσία έχει παρουσιαστεί σε χρόνο ρεκόρ. Το Συμβούλιο χθες υιοθέτησε σχέδιο ε, και σήμερα μετά τη δική σας ψήφιση μαζί με τον πρόεδρο ε, Σούλτς ήδη υπογράψαμε το κείμενο. Και μετά τη δημοσίευση του ε, που θα λάβει η χώρα στις επόμενες εβδομάδες, τα κράτη-μέλη που θα μπορούν να πάρουν την προκατακτική χρηματοδότηση. και η προκαταρκτική χρηματοδότηση θα αυξηθεί στο 1 δις περίπου για το 2015. Δράτω με τις ευκαιρίες λοιπόν να επιβεβαιώσω ότι το Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγες τις εξελίξεις σε σχέση με την κατάσταση της ανεργίας και της απασχόλησης των νέων και του πώς τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και την πρωτοβουλία για την εγγύηση που προσφέρεται στους νέους να έχουμε αποψή μα ότι οι αιτίε πίσω από την ανεργία των νέων είναι πολύ περίπλοκε. Η αυξημένη χρηματοδότηση λειτουργεί συμπληρωματικά με άλλα μέτρα και με άλλε μεταρρυθμίσει που πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν τα διαρθρωτικά ε, προβλήματα που κρύβονται πίσω από την ανεργία των νέων για να μειωθεί η ανεργία ουσιαστικά πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα για να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης. Και τέλος θα ήθελα να τονίσω πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι κοινωνικοί εταίροι σε αυτό το πλαίσιο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσουμε ε, με τις πολιτικές ομάδες. Η κυρία Μογάν Σαχτιέ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω στην εκπρόσωπο του Συμβουλίου απόψε ότι αυτή η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων την ήθελαν τα κράτη-μέλη. Δική τους επινόηση είναι και έκαναν την επικοινωνία επανειλημμένος αυτής της πρωτοβουλίας και θα πρέπει να πω ότι ενίοτε δημιουργήσαν σύγχυση μεταξύ της εγγύησης για τους νέους και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Η δεύτερη ανταποκρίνεται σε πραγματική ανάγκη των πολιτών και μιλήσατε κι εσείς για τη σημασία που έχει ε, για ε, τον αριθμό των νέων ανέργων. Είναι τόσοι πολλοί οι νέοι άνεργοι που θα πρέπει να δράσουμε. Όμως, Κατά την πρώτη ε, χρονιά υλοποίησης ε, ε, υπήρξαν πολλές αδυναμίες. Κάποια καλά παραδείγματα που αναφέρατε δεν υπάρχουν παντού. Για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτέλους λειτουργήσε γρήγορα, εξαιρετικά γρήγορα. Μέσα σε τρεις μήνες από την προκαταρκτική χρηματοδότηση από 1% την πάμε στο 3%. Ευχαριστούμε όλους, όλες τις πολιτικές ομάδες που μας βοήθησαν σε αυτή την αναδρομική ε, εφαρμογή της αύξησης του 1 στα 3%. Ευχαριστούμε τους πάντες, αλλά να ξέρετε ότι δεν θα παρετηθούμε. Θα ε, παρακολουθήσουμε στενά ε, την κατάσταση ώστε να αξιοποιηθούν όλα αυτά τα κονδύλια. Ξέρετε, έχω γνωρίσει πολλούς υπουργούς που συνεχίζουν να μπερδεύουν αυτά τα δύο. Ποια είναι η εγγύηση για τους νέους και ποια είναι η πρωτοβουλία για την απασχόληση για τους νέους. Ε, θέλουμε να υπάρξει καλύτερη επικοινωνία. Βοηθήστε μας, συνεχίσετε να ασκείτε πίεση στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Παρακαλώ, παρακαλώ να μην ξεπερνάτε το χρόνο ε, που σας έχει δοθεί. Ο κύριος Μπενιφέη, Σοσιαλιστές, δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί εκπρόσωποι του Συμβουλίου Μεταχαλάς. Με τα χαρά έχω τη δυνατότητα να ασχοληθούμε με το θέμα τη ανεργία των νέων. Λίγε εβδομάδε πριν την υιοθέτηση του διατάγματο για την αύξηση τη προγραμματοδότηση για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο ζητάμε από το κράτο μέλο να δείξουν σοβαρο... τα κάτι μέλη να δείξουν σοβαρότητα για να θεραπεύσουν την πληγή τη ανεργία των νέων στην Ευρώπη. Θα πρέπει να έχουμε διαβεβαιώσει από το γεγονό ότι το Συμβούλιο είναι διαθεσίμο να πολεμήσει για του νέου του για οποιοδήποτε κόστο do whatever you take», όπως λέμε στα αγγλικά, να χρησιμοποιήσουμε ό,τι χρειάζεται δηλαδή. Το επαναλαμβάνω λοιπόν. Έπεσε, συνεργάστηκε με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινοβούλιο για να τοποποιηθεί ο κανονισμό, επιτρέποντα έτσι την απεμπλοκή των διαφόρων πόρων για τα κράτη σε χρόνο ρεκόρ. Ήρθε η στιγμή όμω τώρα να παραχθούν αποτελέσματα, να ξεκινήσουν τα προγράμματα και να ξεπεραστούν τα εμπόδια δεν πρόκειται μόνο για πρόβλημα οικονομικό. Πάνω απ' όλα θα πρέπει να επιλύσουμε μεγάλα προβλήματα που συνδέονται με υπερβολική γραφειοκρατία όσον αφορά την εγγραφή στα προγράμματα και για του νέου και για τι επιχειρήσει και του εταίρου που θέλουν να συμμετάσχουν. Θα είναι ουσιαστικό να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και την επικοινωνία όσον αφορά αυτά τα προγράμματα να μαθευτούν. Σήμερα είναι ανεπαρκή η προσπάθεια γνωστοποίηση. Πολλοί νέοι, εκείνοι που χρειάζονται περισσότερα προγράμματα, δεν ξέρουν καν ότι υπάρχει αυτή η εγγύηση για του νέου και η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Αυτό είναι παράλογο και θα πρέπει να αλλάξουμε πολύ γρήγορα την προσέγγιση. Θα πρέπει να αυξήσουμε τι προσπάθειε τόσο οι νέοι να έχουν προσφορέ ποιοτικέ και να μην γίνουν ε, κάποιο εργαλείο εκμετάλλευση σε αυτά τα προγράμματα και να μην οδηγήσουν σε επισφαλή εργασία. Θέλουμε λοιπόν να επαγρυπτεί το Κοινοβούλιο και να βοηθά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να ανταποκριθούμε στο ύψο των περιστάσεων που μπορεί να αποφασίσει τη μοίρα μια ολόκληρη γενιά. Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων από μόνη τη δεν σε βαθμό να δημιουργήσει νέε θέσει απασχόληση. Δεν υπάρχουν μαγικέ συνταχηγέ. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι πόλει τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Χρειάζεται και πολιτική ανάπτυξη ταυτόχρονα. Επενδύσει στρατηγικού τομεί και ουσιαστικά χρειάζεται μια πολιτική βιομηχανική ευρωπαϊκή δυνατότητα να το εισόδημα ε, σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση της ανισότητας, ούτως ώστε να έχουμε καλύτερο μέλλον που διασφαλίζουμε για τις μελλοντικές γενιές. Ευχαριστώ. Κύριε Μπενιφέη, διχόσαστε μια γαλάζια κάρτα. Κύριε Μπενιφέη, δέχεστε μια γαλάζια κάρτα. Κύριε Ζάνη, για 30 δευτερόλεπτα ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Βουλευτά που δεχτήκατε την ερώτησή μου. Λοιπόν, και εγώ συμφωνώ και εγώ λέω ότι χρειαζόμαστε πράγματι τη απασχόληση, θέσεις απασχόλησης ποιοτικέ. Αλλά διαβλέπετε να υπάρχει ένα σύστημα αξιολόγησης το οποίο θα είναι επιχειρησιακό, λειτουργικό και έτσι θα έχουμε την εγγύηση ότι οι κυβερνήσεις θα θαπανούν τα χρήματα σε θέσεις εργασίας εικονικές, αλλά ότι η βοήθεια που θα χορηγείται θα έχει πραγματική υπόσταση. Απάντηση. Πιστεύω ότι χρειάζεται ένα κράμα δράσεων. Από τη μία πλευρά μια δυνατότητα αναπτύξης οικονομίας, ούτω ώστε οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται να είναι πραγματικές θέσεις και αυτά, έτσι αυτά τα χρήματα να μην ε, αντικαθιστούν άλλες πολιτικές να ενεργοποιούν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την άλλη πλευρά, με σαφέ ενδείξει και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να επαγρυπνούν ε, τι, και να βλέπουν τι κάνουν τα κράτη-μέλη. Οπότε ε, είναι χρήσιμο γίνονται και τα δύο. Η κυρία Μάκιντάιρ έχει το λόγο για ένα μισή λεπτό. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Η ανεργία στην δική μου χώρα και στην δική μου περιοχή των West Midlands έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Η ανεργία στις ηλικίες 16 έως 24 έχει μειωθεί ταχύτατα το τελευταίο χρόνο. Ωστόσο, τους τελευταίους τρεις μήνες μέχρι το ελάχιστες οι αλλαγές και έτσι είμαστε στο 15,9%. Και τα πιο πρόσφατα στοιχεία του CBI δείχνουν ότι η ανεργία αυξήθηκε τον προηγούμενο μήνα στα δυτικά Midlands. Ό,τι μου και να μας λένε τα στατιστικά στοιχεία, αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι εξακολουθούμε να έχουμε 6.500 νέους από 18 24 χρονών άνεργους στην πόλη του Birmingham. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι είναι επιτυχές και τι όχι. Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων έχει αποφέρει πολύ λιγότερα από όσα προσδοκούσαμε και πιστεύω ότι είναι πολύ ανησυχητική η έκθεση τρικτικού συνεδρίου. Και καλωσορίζω την ευκαιρία ανταλλαγή απόψεων με την Ελιάνα Ιβάνοβα στην Επιτροπή απασχόληση στην σχετική ειδική έκθεση. Γιατί αν ε, δεν είναι θετικό ο αντικτύπο της ε, πρωτοβουλία απασχόληση των νέων, θα πρέπει να εξετάσουμε τα αίτια τη αποτυχία αυτή. Θα κοιτάξουμε την ε, άλλη εβδομάδα και το πακέτο της νομοθεσίας. Και όπως είπε ο κύριος Τίμερμανς, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί από εκεί θα έρθουν ε, οι δουλειέ και για τους νέους. Η κυρία Χάρκιν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητό Συμβούλιο. Είμαστε εδώ για να θέσουμε ερωτήματα για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Κάποια ερωτήματα έχουν ήδη τεθεί. Γιατί ήταν τόσο μικρή και, και αργή η απορροφικότητα, γιατί υπήρξε αυτή η καθυστέρηση και πότε μπορούμε να, περιμένουμε βελτίωση. Δεν χρειάζεται να σας επαναλάβω τα στοιχεία γιατί τα ποσοστά ανεργία των νέων όλοι τα ξέρουμε και είναι παράδεκτα υψηλά. Θέλουμε με την πρωτοβουλία αυτή να προσθέσουμε αξία στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, μέχρι τώρα δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη επιπρόσθετη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να υπάρχει επιτυχία, το Συμβούλιο θα πρέπει να διδραματίσει το ρόλο του. Είναι κρίσιμο για την εφαρμογή τη πρωτοβουλία εφαρμογή, πρωτοβουλία απασχόληση των νέων. Υπάρχουν πολλέ ευκαιρίε για μαθητείε, για την ε, πρώτη απασχόληση επιδοτήσεις για την απασχόληση, μέτρα για την εκπαίδευση, για την κινητικότητα, για τους νέους επιχειρηματίες. Το Συμβουλίο μας έχει πει ήδη ότι η πρωτοβουλία και η εγγύηση για απασχόληση των νέων δεν είναι πανάκια. Το ξέρουμε αυτό, αλλά είναι σημαντικά μέτρα σε έκταση και το θέμα αυτό μας απασχολεί ιδιαίτερα. Όπως αναφερθήκε και στην προφορική ερώτηση, θέλουμε γρήγορη αποτελεσματική εφαρμογή της προχρηματοδότησης με τα σωστά αποτέλεσματα. Η συνάδελφος κ. Μακιντάρ έθεσε το θέμα της έκθεσης του ελεκτικού συνεδρίου. Είχαμε ήδη ανταλλαγή απόψεων με το ελεκτικό συνεδρίο και κάποια θέματα θα πρέπει να επιληθούν. Το γεγονός ότι δεν έγινε εξάντα αξιολόγηση, ότι τα κράτη-μέλη δεν έδωσαν επαρκείς πληροφορίες για τη χρηματοδότηση σε ό,τι αφορά το σχέδιο εφαρμογής της πρωτοβουλίας. Τα θέματα αυτά θα πρέπει να επιληθούν, αλλά θέλουμε τα κρατημέλη ουσιαστικά να αναλάβουν τις ευθύνες τους και άμεσα να εφαρμόσουν την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Ευχαριστώ. Για λεπτό, κυρία από την ε, Πέρα από τις λογικές αμφιβολίες που βρίσκονται στην ερώτηση της Μαρίτα Ολκούχ, υπάρχει και ένα δομικό πρόβλημα. Η πολιτική των περικοπών κάνουν τις χώρες που τις εφαρμόζουν ουσιαστικά να έχουν ως μοντέλο νορμάλ την αβεβαιότητα. Να δουλεύει κανείς και να μην τα βγάζει πέρα μέχρι το τέλος του μήνα. Για να δημιουργήσουμε απασχόληση πρέπει να βρούμε μια λογική λύση στο πρόβλημα του χρέους στην Νότια Ευρώπη, να εκδημοκρατήσουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να γίνει μια προοδευτική φορολογική μεταρρύθμιση που θα κάνει τους πλούσιους να πληρώνουν περισσότερους φόρους. Ε, εν μεταξύ και μέχρι να τα καταφέρουμε αυτές οι πρωτοβουλίες για τις οποίες μιλάτε είναι μια, ένα πρόσχημα έτσι ώστε δημόσια κονδύλια να πηγαίνουν σε ιδιωτικέ επιχειρήσεις και ξεκινούνται από ένα, ξεκινούν από ένα, μια εσφαλμένη παραδοχή ότι δηλαδή οι νέοι δεν είναι απασχολήσιμοι, ότι αυτοί δεν, είναι, δεν έχουν απασχολησιμότητα. Η νεανική αυτοαποσχόληση ουσιαστικά οδηγεί σε υπερχρέωση και σε χρεοκοπία. Μπαίνουν σε μια αγορά που δεν υπάρχει ούτε αγορά ούτε καταναλωτές. Η ζήτηση και αγορά και οι υπηρεσίες που μπορούν να δώσουν συνεταιρισμοί θα συρρυκνούνται όλο και περισσότερο. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν ότι το αίτημα μας είναι μια νέα οικονομική πορεία ε, με στόχο τη δημιουργία χρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης. Ευχαριστώ. Η κυρία και από τους Πράσινους για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί εκπρόσωποι του Συμβουλίου, σήμερα συζητούμε διότι η Επιτροπή για την Κοινωνική Απασχόληση έχει υιοθετήσει ένα κείμενο για την πρωτοβουλία για την απασχόληση για τους νέους και την εφαρμογή του από, από τα κράτη-μέλη. Το 99% των πολιτών δεν έχουν ιδέα περί τίνος πρόκειται αυτή η συζήτηση. Καλύτερο λοιπόν να το εξηγήσω. Στο ερώτημά μας λέγεται ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει κάνει την ανεργία των νέων να φτάσει σε αστρονομικά επίπεδα στα κράτη-μέλη. Και να σας το μεταφράσω αλλιώς αυτό. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές μετά την απορρίθμιση της ατζέντα, το μόνο που έκαναν ήταν να διαλύσουν τις αγορές εργασίας τα τελευταία χρόνια και η πληθυσμιακή ομάδα και η κοινωνική ομάδα που επλήγει περισσότερο είναι οι νέοι. Είναι κοινό το μοντέλο που χρησιμοποιείται. Ε, καταδικάζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία αντιδρά και δίνει κάποια χρήματα. Λίγα, αλλά εν πάση πτώση δίνει χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταπολεμήσει την ανεργία των νέων και τα χρήματα πρέπει να τα ξοδέψουν τα κράτη-μέλη στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία των νέων. Τα αποτελέσματα επί τόπου λοιπόν δεν ανταποκρίνονται στις αρχικές προσδοκίες λέγεται στο κείμενο wow έχω να πω είναι εξαιρετικά διπλωματική και δεν μπορεί καν να μεταφραστεί αυτή η πρόταση γιατί ξέρετε πάρα πολλοί θεωρούν εξωφρενικό το γεγονός ότι τα χρήματα που δίδονται στα κρατημέλη για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων δεν έχουν απορροφηθεί επαρκώς μετά από 22 μήνες και ε, ως κοινοβουλευτική έχουμε αυτή την προφορική ερώτηση για να πούμε στα κρατημέλα Κρέτη μελη ξεκάθαρα ότι επιτέλους πρέπει να δράσουν τώρα. Και ελπίζω πολλοί πολίτες να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα, να βγουν στους δρόμους, να πλημμυρίσουν τους κυβερνώντες τους με επιστολές, καλώντας τους να αναλάβουν δράση. Από η FTD, κυρία Ατζέα, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την εκπρόσωπο του Συμβουλίου, ευχαριστώ τους συναδέλφους. Εγώ επανειλημμένα διερωτήθηκα γιατί τέτοια ανεπάρκεια, γιατί τόσο προφανής ανεπάρκεια όσον αφορά μια πρωτοβουλία που έπρεπε να έχει ακριβή σκοπό και στόχο, αλίμονο η πύληση του προβλήματος της ανεργίας δεν είναι η αύξηση της ανεργίας. Δυστυχώς μέχρι τώρα εργαζόμαστε για την εμετώπιση σοβαρότητα του προβλήματος ανεργίας δεν μας επιτρέπει το πρόβλημα να έχουμε αποκοπόθεσμα σχέδια. Δεν μας επιτρέπει που δεν είναι να σκεφτούμε το μέλλον, να δημιουργήσουμε απασχόληση και να καινοτομούμε. Η συνάδελφος Μωρέν Σαχτιέ έκανε μια διευκρίνηση. Είπε συχνά συγχαίωμε την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων με την εγγύηση για τους νέους. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που συχνά έχουν οι υπουργοί και αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Πολύ συχνά, δυστυχώς, είμαι υποχρεωμένη να πω ότι πιθανότατα δεν γνωρίζουν καν ποια είναι η πρωτοβουλία για την ανεργία των νέων και δεν ξέρουν εξίσου ποια είναι η εγγύηση για τους νέους και δεν μπορούν να κάνουν τη διαφοροποίηση μεταξύ των δύο και να αποφασίζουν τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο. Αυτό είναι ακόμα σοβαρότερο, διότι αν εγνώριζαν τις ευκαιρίες που δημιουργούνται, θα ετοίμαζαν ειδικά προγράμματα που θα λάβανα πραγματικά υπόψη τις απαιτήσει των νέων, τις ανάγκες τους. Εάν γινόταν αυτό, πιθανότατα θα μπορούσαμε να έχουμε πολιτικές πολύ αποτελεσματικότερες, κάτι που δυστυχώς στη χώρα μου δεν έγινε. Χάσαμε όλους τους στόχους. Θα μπορούσα να ρωτήσω κάτι. Διότι εξακολουθώ να ντρέπομαι για τον τρόπο με τον οποίο σπαταλώνται οι ευκαιρίε που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάντε ένα προσεκτικό έλεγχο. Πώ χρησιμοποιούνται αυτοί οι πόροι από τι χώρε και από τα κράτη-μέλη. Πρέπει να επαγρυπνείτε, να αγρυπνείτε, να ελέγχετε τα προγράμματα, του τρόπους εφαρμογής τους. Ελέγχετε πού και πώς αυτά τα χρήματα, διότι σας εγγυώμαι ότι οι νέοι που ε, βοηθήθηκαν από αυτά τα προγράμματα μετρούνται στο δάχτυλο, στα δάχτυλα του ενό χεριού. Αυτή είναι η πραγματικότητα και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ζητείτε έλεγχο, παρακολούθηση, προσεκτικό έλεγχο και συνεχής. Πώ χρησιμοποιούνται αυτά τα χρήματα. σα ευχαριστώ. Δεν βλέπω τον κύριο Φουντούλη. Θα πάμε στην κυρία Λόπε Φοντανιέ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν θεωρούσα ότι θα πάραμε στο λόγο. Θα ήθελα να πω ότι τα αποτελέσματα που έχουμε πετύχει δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες μας και γι' αυτό πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί έτσι ώστε η πρωτοβουλία να είναι χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο. Ένα από τα βασικά εμπόδια φαίνεται να έχει λυθεί. Η εφαρμογή της προκαταρκτικής της έγκαιρης ε, χρηματοδότησης θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη που δεν μπορούσαν να βάλουν τα ίδια ε, τα κονδύλια λόγω έλλειψης ρευστότητας να μπορούν να ε, κάνουν τα απαραίτητα βήματα έτσι ώστε οι νέοι να προσχωρήσουν στην αγορά αγορά και θα πρέπει να είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε και άλλα εμπόδια για να τα καταρρύψουμε. Ε, είμαι αισιόδοξη. Επιτρέψτε μου να παρουσιάσω το παράδειγμα της δικής μου χώρας. Η Ισπανία είναι μία από τις χώρες όπου η ανεργία των νέων έχει εκτοξευθεί. Έχει αποκεντρωμένο ε, μοντέλο το οποίο επιβραδύνει την ε, εφαρμογή αυτή, αυτού του εργαλείου. Παρόλα στις αντικσοότητες ήμασταν από τους πρώτους που αξιοποιήσαμε αυτό το εργαλείο. 43% ε, των εγγραφών σε αυτό ε, το, των δικαιούχων είναι γυναίκες. Έχουμε πάρα πολλές εκστρατείες επικοινωνιακές οι οποίες ε, αυξάνουν εκθετικά τον αριθμό των συμμετεχόντων. Ήδη έχουμε φτάσει στους 40.000. Τα εμπορικά επιμελητήρια μπορούν να συμβάλλουν περισσότερο, οι επιχειρήσεις επίσης, αλλά και οι σύμβουλοι, οι εταιρείε συμβουλευτικής αναζήτησης εργασίας για την επίτευξη των στόχων. Αυτά ευχαριστώ. Η κυρία Στάινρουκ για ένα λεπτό. Είναι λυπηρό πόσο πολύ καιρό διαρκεί και πόσο καταρακώνονται οι ευκαιρίες πολλών νέων λόγω του αντιεξόδου. Αλλά δεν θα σταματήσουμε εδώ στο Κοινοβούλιο να πολεμάμε για την καταπολέμηση της ενέργειας των νέων και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό που τίθεται το ερώτημα αυτό το προφορικό σήμερα προς το Συμβούλιο. Γιατί η ανεργία των νέων και η μείωση της, η μηδενική ανεργία των νέων είναι κάτι από το οποίο απέχουμε φωτός. Ε, ωραία λόγια, ωραίες ε, σύνοδοι, ωραίες υποσχέσεις, αλλά τίποτα δεν πραγματοποιείται και πάντα ανακύπτουν ε, τι και δικαιολογίε για την αποτυχία. Μία δεν υπάρχουν χρήματα και όταν υπάρχουν χρήματα δεν υπήρχε προχρηματοδότηση. Και αυτό το λύσαμε λοιπόν ως πρόβλημα και τώρα... Τώρα επιτέλους δεν πρέπει να υπάρξουν άλλες δικαιολογίε. Τα κράτη-μέλη τώρα θα πρέπει πραγματικά να δράσουν και να υπάρξουν ορατές πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν τους νέους. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα η κυρία Ζητνάσκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ξέρουμε ότι η αρχική πρόταση αύξησης της προσχηματοδότησης έχει λάβει εμβρία υποστήριξη εδώ στο Κοινοβούλιο, αλλά δεν πρόκειται για μια λευκή επιταγή. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τις δικαιολογίε για το τι, ποιε είναι οι αιτίε που αποτυγχάνει το πρόγραμμα. Το θέμα είναι οι νέοι να ωφεληθούν από τα προγράμματα, αλλά στη Φιλανδία η ενεργοποίηση των ε, νέων ανέργων έχει πετύχει, ενώ χάρη στις χώρες που ε, αντιμετωπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα, αυτό σημαίνει ότι κάτι θα πρέπει να αλλάξει στη μέθοδο. Γι' αυτό λοιπόν με ενδιαφέρε η απάντηση του Συμβουλίου. Αν ε, παρά την αύξηση των πόρων δεν μπορούν τα κράτη-μέλη να βοηθήσουν τους νέους, μήπως υπάρχουν άλλοι τρόποι για να βοηθήσουμε καλύτερα τους νέους. Κυρία Γκλαμπάγεβα, για λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία εκπρόσωπε του Συμβουλίου, η πρωτοβουλία για την ενεργεία των νέων, πέρα από μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, είναι ένα από τα κρίσιμα εργαλεία για την βελτίωση της ζωής των νέων. Γι' αυτό πιστεύω ότι τα 1,2 τα παραπάνω ευρώ που διατίθενται είναι όλος ιδιαίτερο σημαντικά και χαίρομαι πάρα πολύ που εγκρίθηκε το ποσό σε χρόνο ρεκόρ. Αποτελεσματική συνεργασία, λογική συνεργασία είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε τους νέους. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαφορέ όσον αφορά τα επίπεδα ενεργεία μεταξύ των κρατών μελών. Υπάρχουν τεράστιε διαφορέ. Υπάρχουν χώρε όπου υπάρχουν περισσότεροι άνεργοι νέοι από ό,τι απασχολούμενοι νέοι. Άλλε χώρε όμω τα πάνε τόσο καλά που δεν είναι καν επιλέξιμε για τα μέτρα αυτά. Ελπίζαμε ότι η εμπροστοβαρής προσέγγιση θα προωθούσε την ταχύτερη εφαρμογή των μέτρων. Τώρα εκπλησόμεθα διότι βλέπουμε ότι δεν απορροφώνται τα ποσά. Είναι προβλήματα διοικητικά, υπάρχουν διοικητικά εμπόδια, υπάρχουν αόριστοι ορισμοί όσον αφορά την ποιοτική θέση απασχόλησης, υπάρχει αοριστία ε, και έτσι και οι στόχοι είναι αόριστοι. Η πρωτοβουλία υποτίθεται ότι συμβάλλει στην αλλαγή της καταστάσεως της αγοράς εργασίας. Εσείς πώς θα προσπαθήσετε να δώσετε τα κίνητρα στα κάτι μέλη να κάνουν περισσότερα για αυτό το σκοπό. κυρία Ντελή, έχω ένα μήνυμα πάρα πολύ εύκολο να σας διαβιβάσω πείτε σε αυτού του κυρίου, του αρχηγού κρατών κυβερνήσεων, σταματήστε τον μπλα μπλα, εστέ τολμηροί, αποδείξτε ότι έχετε θάρρο. φροντίστε ούτω ώστε προτεραιότητα των πολιτικών επιλογών σα είναι η απασχόληση των νέων. Μέχρι τώρα είναι ντροπή. Σύμφωνα με το ελεκτικό συνέδριο, καμιά θέση απασχόληση δεν δημιουργήθηκε χάρη στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Νεολαία. Λοιπόν, τα κράτη-μέλη φταίνε και δεν δικαιολογούνται διότι αυξήθηκε και το ποσό που ετίθεται. Χρειάζεται η βελτίωση του διοικητικού ε, μηχανισμού για να ειδοποιηθούν και να κινητοποιηθούν οι νέοι. Πρέπει να οικοδομήσουμε το μέλλον. Έχει γίνει κρατών κυβερνήσεων που καταλάβουν ότι ότι οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, γεωθερμικέ πηγέ ενέργεια είναι το μέλλον. Ψηφιακό τομέα. Εκεί χρειάζονται επενδύσει. Γιατί? Διότι όλοι αυτοί οι τομεί δημιουργούν θέσει εργασία βιώσιμε που δεν μετεγκαθίστανται. Κύριοι αρχηγοί κατών και κυβερνήσεων, και κλείνω εδώ. Μέχρι τώρα δεν έχετε πλέον δικαίωμα να κάνετε ανακοινώσει. Και η νεολαία δεν είναι απλώ μια μεταβλητή προσαρμογή. Ευχαριστώ. Ο κύριο Άρνοτ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ποιο θα μπορούσε να μαντέψει ότι θα καταλήγαμε εδώ μια τέτοια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που δεν έχει αποδώσει πόρους και αποτελέσματα. Μια μεγάλα ιδέα για την ε, κατασπατάληση των ε, χρημάτων των φορολογουμένων με απογοητευτικά αποτελέσματα και θα καταλάβουν τα κράτη-μέλη ότι αυτό που προσπαθεί να κάνει το Κοινοβούλιο είναι να τους επιβάλλει πράγματα Υπάρχουν απλά συναλλακτικέ λήξει. Οι Βρετανοί, φορολογούμενοι για βρετανικά έργα, για βρετανού ανέργου. οι Γερμανοί, για Γερμαν... Γερμανοί φορολογούμενοι για γερμανικά project, οι Λετωνοί για τα λετωνικά project. Είναι τόσο απλό και ξεκάθαρο. Δεν χρειάζεται να επικρατήσει ο τρόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σταματήστε να παρεμβαίνετε. Αφήστε τις χώρες να τα πανάνε τα δικά τους χρήματα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε τη Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόληση, πολύ συχνά θέσατε το τελευταίο ερώτημα. Τι πρέπει να κάνουμε αν η αύξηση τη προχρηματοδότηση δεν έχει κανένα αντίκτυπο σε 12 μήνε. Σίγουρα υπήρξε έλλειψη διάβγε. δεν υπήρχε καλή σχέση αιτίου και αιτιατού. Δεν χρησιμοποιήθηκαν σωστά οι πόροι ευρωπαϊκοί για την ανακούφιση ανεργία των ε, νέων. Δεν μειώνεται η ανεργία. Έχουμε περισσότερη ανεργία, αλλά μεγαλύτερο φόρτο όσον αφορά τα κοινωνικά επιδόματα, λιγότερη απασχόληση, ένα φαύλο κύκλο που ξέρουν τα κράτη-μέλη. Πρέπει να φύγουμε από τα λόγια και την ορολογία που χρησιμοποιούνται 30 χρόνια στα θεσμικά όργανα και περάσουμε στι πράξει. Θα αφήσουμε στι επιχειρήσει να κινηθούν σε κάτι μέλη, τι μικρομεσαίε κυρίω, να απελευθέρωσουμε του περιορισμού του νομικού για την επαγγελματική κατάρτιση, για την απασχόληση, να αρθούν οι τροχοπέδοι, ε, οι όσον αφορά την εκπαίδευση. Θα πρέπει λοιπόν, ε, θα πρέπει σε ένα χρόνο και εκτό εκπλήξεω πιστεύω ότι τα αρνητικά αποτελέσματα εκ των προτέρων θα είναι γνωστά αν δεν αλλάξουν όλα αυτά. Η κυρία Γιονγκέριους έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχει έρθει και το καλοκαίρι. Και έχουμε κλείσει 8 χρόνια περίπου από τότε που μας χτύπησε η μεγάλη οικονομική κρίση στην Ευρώπη. Οι τράπεζες, ε, η ανεργία αυξήθηκε και έξι ε, γενιές έχουν βγει στην αγορά εργασίας ε, με τέτοιες φτωχές συνθήκε και παντού είναι πολύ υψηλή η ενέργεια των νέων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητήσε μια νέα προοπτική για τους νέους στις πιο πληττόμενες περιοχές και πλέον υπάρχουν χρήματα στην προγραμματοδότηση, προγράμματα για να υποστηρίξουν τους νέους στην αγορά εργασία για να μην περιμένουν από τις κυβερνήσεις τους για τη συγχρηματοδότηση. Δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο αλλά είναι καταπήγουσα η ανάγκη. Σε έξι μήνες θα πρέπει να ξέρουμε κατά πόσο βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε οκτώ ε, φουρνιές ε, από φύτων χωρίς προοπτική στην αγορά εργασία. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό το λόγο έχει και ο Κλειβέζης. Ο κύριος Καλβέ Τσαμπών. Κυρίες και κύριοι, εάν ε, Υπάρχει ένα πράγμα που πραγματικά θέτει σε κίνδυνο την αξιοπιστία της Ευρώπης και του ευρωπαϊκού οράματος, του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, ε, τότε αυτό είναι η μαζική ανεργία των νέων. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χάσει την αξιοπιστία της αν χάσει αυτή τη μάχη. Πολύ καλά είναι όλα αυτά που λέτε, Ας κάνετε ό,τι νομίζετε, να πάτε να δουλέψετε στα κράτη-μέλη. Να μην παρουσιάζουν άχρηστες δικαιολογίε τα κράτη-μέλη, ότι δηλαδή υπάρχει διοικητική αποκέντρωση, ότι δεν έχουν αρκετή εξουσία, ότι τα χρήματα τους φτάνουν καθυστερημένα και ούτω καθεξής. Η εκάστοτε κεντρική κυβέρνηση αυτά λέει. Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά είναι αστεία παράδοξα όλα αυτά που γίνονται. Πρέπει κάτι να γίνει για να μπουν οι νέοι στην αγορά εργασίας και μάλιστα χθες, όχι σήμερα. Ο κύριος Λόπες, για ένα λεπτό παρακαλώ. Εκτός μικροφώνου μιλητής. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι δεν έχουμε αξιοποιήσει πλήρως αυτή την πρωτοβουλία ακόμα. Κάναμε προσπάθεια για την προκαταρκτική, την έγκαιρη χρηματοδότηση των κράπο, στα κράτη-μέλη. 5 ε, εκατομμύρια είναι οι νέοι άνεργοι που είναι κάτω των 25 ετών στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Το Ευρωβαρόμετρο προ λίγο μας υπενθύμησε ότι μόνο 8 στους, σε κάθε 10, 8 στους 10 έχουν ακούσει να γίνεται λόγος για αυτή την πρωτοβουλία. Η Ισπανία είναι σημαντική, θα παρουσιάσει το παράδειγμά τη, όχι μόνο γιατί η ανεργία των νέων είναι πολύ μεγάλη, αλλά διότι είναι η πρώτη χώρα σε πόρους. 800 νέοι άνεργοι έχουν δηλωθεί δεν έχουν βρει δουλειά ούτε ε, ακολουθούν κατάρτιση και έχουμε και μειώσεις γίνονται διάφορα σκανδαλώδη πράγματα. Απολύουν τον πατέρα κάποιου για να τον προσλάβουν τον νέον με τα μισά λεφτά. Είναι σκανδαλώδη όλα αυτά να αναφέρω κάποιε ανησυχίε για το πώ χρησιμοποιούνται τα χρήματα αυτά στι κράτη-μέλη για την αξιολόγηση αντικτή που Χρειάζονται κάποια κριτήρια. Και η ενίσχυση για την ανεργία των νέων είναι ένα από τα κριτήρια στην Ανατολική και Νότια Ευρώπη. Βλέπουμε ταχύε αλλαγέ όσον αφορά τον νέο πληθυσμό λόγω μετανάστευση. Παραδείγματο χάρη, το επίπεδο τη ανεργία στην Εστονία μειώθηκε από 17% που ήταν στην αρχή σε περίπου 12% το τέλο του 2014. Τι επιτυχία φαίνεται αυτή. Αλλά αν μειώνεται η ανεργία είναι γιατί φεύγουν οι νέοι. Και αυτό δεν δείχνει ότι είναι αποτελεσματικά τα το προβλήματα και κοινωνικέ ομάδε έχουν μεγάλη ενεργεία στη χώρα μου. Ετήσιο επίπεδο ενεργεία για του εθνοτικού Εστονού είναι 1,6 ε, φορέ λιγότερο από του ρωσόφωνου. Και είναι 27% οι ρωσόφωνοι σε αυτή την ομάδα. Αλλά η ενεργεία του είναι 21%. Τα στατιστικά στοιχεία, τα μη ομοδοποιημένα, είναι κρίσιμη σημασία για τη σωστή ανάλυση των μέτρων συμπεριλαμβανομένου και του μέτρου αυτού τη εγγύηση για του νέου. Ευχαριστώ. Ο κύριο Πάβελ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα... θα ήθελα να ξεκινήσω καλωσορίζοντας ε, την απόφαση να αυξηθεί η προγραμματοδότηση της ε, πρωτοβουλίας απασχόλησης των ε, νέων για να υπάρξει ο μεγαλύτερος δυνατός αντίκτυπος καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αφιερώσει όσο πιο πολλά κονδύλια γίνεται για την πρόθεση της απασχόλησης των νέων και των γυναικών και νομίζω ότι θα πρέπει να συνεργαστεί και με το Ευρωπαϊκό με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να υπάρξουν μηχανισμοί χρηματοδότησης για επιχειρήσεις, για νέους επιχειρηματίες και γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να υπάρξει η ανάπτυξη, για να υπάρξει αυτή η δημιουργική δύναμη που θα παραμείνει στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά θέματα εκπαίδευση. Θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και πρακτικοί και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν πιο εντατικά με τους βασικούς φορείς, ε, τις κυβερνήσεις, τους ε, εταιρείε, του εργοδότες, ε, τους υπεύθυνους εκπαίδευσης και με τις ε, οργανώσεις ε, της κοινωνίας των πολιτών σε κάθε κρατός μέλος. Ως εκπρόσωπος της νέας γενιάς πιστεύω ότι το σχολείο θα πρέπει να δίνει πραγματικά παράθυρα για το άνοιγμα στην αγορά εργασία. Ο κύριος Σάιμον για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αυτό το όλο σχήμα λειτουργούσε για ένα χρόνο πριν τον Μάρτιο του 2014 η συντηρητική κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν παρουσίασε προγράμματα για να αντλήσει χρήματα. Και τότε μόνο πρότειναν να πάρουν ελάχιστα ποσά. 206 εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα για να βοηθήσουν οι νέοι στην περιοχή μου στα Δυτικά Μίτλαντς να ξαναβρούν δουλειά. Και το Ηνωμένο Βασίλειο, η κυβέρνησή του με τους συντηρητικούς δεν έκανε καμία πρόταση για να αντλήσει τα χρήματα. Και κινήθηκε και ένα χρόνο αργότερα. Και αρνήθηκε να δεχθεί τους βασικούς κανόνες που ισχύουν για όλους τους άλλους στην Ένωση. Για να μπορέσουν να αντληθούν τα χρήματα. Δεν πήραν καθόλου χρήματα και δεν παίρνουν τα χρήματα αν δεν ακολουθήσουν το δικό τους ιδιαίτερο τρόπο. Αποτέλεσμα, οι νέοι στα δυτικά Midlands ε, δεκάδες χιλιάδες από αυτούς παραμένουν άνεργοι. Ο κύριος Πυρίνσκι έχει το λόγο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι το εξής. Ποια είναι η στάση του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της εγγύησης των νέων που έχει επί σειρά ετών ε, προωθηθεί έντονα. Έχουμε θέσει μια προφορική ερώτηση η οποία και δεν απαντήθηκε. Επιτρέψτε μου να επαναφέρω κάποια στοιχεία στη συζήτηση. Το Συμβούλιο θα δεσμευθεί για να ξεκινήσει την εφαρμογή έξι μήνες μετά την θέση σε εφαρμογή της εγγύησης για τους νέους. Και τι προτίθεται να κάνει το Συμβούλιο σε περίπτωση που προκύψει ότι η εγγύηση για τους νέους δεν οδηγήσει σε οποιοδήποτε το αποτέλεσμα. Αυτά τα ερωτήματα είναι δύο από τα πιο σημαντικά ζητήματα. Και πιστεύουμε ότι σε κάθε Συμβούλιο Επασχόληση θα πρέπει να το θέμα αυτό. 135 δισεκατομμύρια ε, ευρώ ανά έτος. Το ξέρετε αυτό το, αριθμητικό στοιχείο, τόσο κοστίζει η ενέργεια των νέων κάθε χρόνο. Παρά όλα αυτά, σε πολλές χώρες υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την απορρόφηση των κονδυλίων. Και οι νέοι ήδη επικρίνουν το πρόγραμμα αυτό. Γιατί δεν φτάνουν τα μέσα αυτά στους νέους τελικά. Αξιότομοι εκπρόσωπε, του Συμβουλίου. Θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή σε μια εκστρατεία των συνδικάτων ε, των νέων «Back to our future». Αυτή η εκστρατεία καταδεικνύει με σαφήνεια την εικόνα που υπάρχει στους, μεταξύ των νέων. Για την διάσωση των ε, τραπεζών ε, διαθέσαμε υπέρογκα ποσά, αλλά για την διάσωση των νέων τα ποσά αυτά είναι ανεπαρκή και φτάνουν πολύ αργά. Ελπίζω ότι όλα τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να υποστηρίξουν την ε, τοποθέτηση που υποστηρίζει και το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μάνι, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Όλοι μας αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε 5 εκατομμύρια νέους που δεν έχουν δουλειά και δεν έχουν προοπτική. Δεν θέλουμε να τους παρηγορήσουμε με όμορφα λόγια. Θέλουμε συγκεκριμένα μέτρα η ευρωπαϊκή λοιπόν εγγύηση αλλά και η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. 6 δις ευρώ. Πιο πολλά θα πρέπει να δούμε. Αν δεν λειτουργούν όμως οι περιφέρειες και οι δήμοι για τις αρμοδιότητες, αν δεν φτάνει η βασική χρηματοδότηση, το μόνο που κάνουμε είναι να αποτρέπουμε τους υπεύθυνους φορείς από την επαρκή δράση. Γι' αυτό λοιπόν θα εφαρμοστεί καλύτερα η πρωτοβουλία για τους νέους αν αυξηθεί η προσματοδότηση από 1 σε 3%. Ας φροντίσουμε να συμμετάσχουν στη διαδικασία στο Συμβούλιο και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν θέλουμε να αφήσουμε μόνους τους, τους ε, όσους πλήττονται. Αυτό το μήνυμα θέλουμε να διαβιβάσουμε. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Κούπουλα Νάτρη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρία εκπρόσωπε του Συμβουλίου, η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων ήταν άκρος ευπρόσδεκτη όταν προτάθηκε το 2013. Έγινε πολλής λόγος για το μέτρο αυτό. Θεωρήθηκε ότι έτσι δείχναμε ότι εδώ είναι η για τους νέους. Όμως οι υποσχέσεις ήταν πολύ μεγάλες. Τα χρήματα όμως δεν έφτασαν στους νέους. Δεν θα πρέπει να παρετηθούμε από τις προσπάθειές μας. Πρέπει να βρούμε νέες μεθόδους να βοηθήσουμε τους νέους. Η μέθοδός μας θα πρέπει να είναι τέτοια που να βοηθάει τους νέους. Θα πρέπει να κινητοποιηθούν επιχειρήσεις, οι ενώσεις των νέων. Και υπάρχουν και διάφοροι άλλοι τομείς που μπορούμε να βοηθήσουμε με πιο ήπιο τρόπο. Δεν είναι θέμα που αφορά τη νέα γενιά και μόνο. Πρέπει να βοηθήσουμε τους νέους να έχουν τη δυνατότητα να έχουν κατάρτιση και μαθητεία για να μπορέσουν να προθηθούν. Πάμε στις παρεμβάσεις κατόπιν ετήματος. Οκτώ έχω στον κατάλογό μου. Η κυρία Ριμπέρο είναι η πρώτη. Θα πάρει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο χρόνια έχουν περάσει από την έναξη της πρωτοβουλίας και δεν υπάρχουν οι καρποί που περιμέναμε, κοιτώντας την ανεργία των νέων, είναι ακόμα σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα, ενώ υπάρχουν ουσιαστικά δυνατότητες πλέον για την απορρόφηση των πόρων. Θα πρέπει να ζητήσουμε από το Συμβούλιο να καταλήξει σε μια γρήγορη απόφαση. Θα πρέπει να κοιτάξουμε και να ακολουθήσουμε και το παράδειγμα της Πορτογαλίας. Ε, λάβαμε προγράμματα λιτότητας αυστηρής λιτότητας και είχαμε πολύ υψηλή ενεργεία νέων, αλλά βλέπουμε ότι η πολιτική αυτή αποδίδει καρπού στην Πορτογαλία. Έχουμε και την, ε, την εγγύηση για τους νέους που έχει βοηθήσει πάρα πολλούς νέους. Είναι 2,2% η μείωση στην ενεργεία των νέων οι νέοι κατά από 25 ετών ωφελούνται και έτσι λοιπόν μειώνεται η ανεργία μεταξύ των νέων. 6 εκατομμύρια νέοι είναι άνεργοι. Και αυτό δημιουργεί ερώτημα για μας. Πώς μπορεί η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων να δημιουργήσει θέσεις εργασίας κυρίως για τους πλέον μειονοκτούντες, παρόλο που αυξήθηκε η προχρηματοδότηση. Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι προβληματική, θα πρέπει να κινητοποιηθούν τα κράτη-μέλη. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να δημιουργηθούν προγράμματα μέσω των χρημάτων. Θα πρέπει να δίνουμε χορηγίες σε σχολεία, σε επιχειρήσεις, βάσει του κανόνα de να αποφευθεί εθνική γραφειοκρατία. Χρειαζόμαστε εύχριστα προσβάσιμα μέτρα. Κάθε μέρα που περνάει είναι μια μέρα χαμένη. Έχουμε πολλά εκατομμύρια νέων που έχουν χάσει την ελπίδα και θα πρέπει να τους δώσουμε κάτι, να κάνουμε κάτι για αυτούς. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Η λιτότητα έχει γεμίσει στρατιές ανέργων την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πάνω από 5 εκατομμύρια άνεργους νέους. Στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2014 το ποσοστό ανεργίας ήταν 50,5% τον ιανουάριο του δύο στην ιταλία το ποσοστό ανεργίας των νέων 41,5%, στην ισπανία. 50,9%. αν θέλουμε πραγματικά να χτυπηθεί η ανεργία των νέων πρέπει να αλλάξουμε πολιτική πρέπει να σταματήσει η πολιτική της λιτότητας πρέπει να γίνει διαγραφή του του χρέους. δεύτερον πόσο είναι το ποσό το οποίο διατίθεται για να στηρίξουμε την απασχόληση των νέων έξι δισεκατομμύρια ευρώ για την πρωτοβουλία για την απασχόληση δέκα δισεκατομμύρια ευρώ για την εγγύηση για την νεολαία. ο κύριος ντράγκη διαθέτει ένα ένα τρισεκατομμύρια ευρώ για την ποσοτική χαλάρωση. και τέλο ξέρετε γιατί δεν αποδίδουν τα μέτρα αυτά; διότι χρειάζεται κρατική συγχρηματοδότηση τα κράτη μέλη δεν διαθέτουν τα κεφάλαια αυτά. στην ελλάδα πρέπει να διατεθούν 160 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό κράτος για συγχρηματοδότηση της πρωτοβουλίας που θα είναι 160 επίσης εκατομμύρια ευρώ από την ευρωπαϊκή ένωση. ευχαριστώ. Πρέπει να σέβεστε το χρόνο κυρία Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, τα 60 δευτερόλεπτα που έχω σήμερα θα τα αξιοποιήσω όχι για να καταδείξω προβλήματα, αλλά για να αναδείξω λύσεις. Αν θέλετε λύσεις για το πρόβλημα της ανεργίας των νέων, θα πρέπει να έχουμε ε, χρήσιμη προσέγγιση. Δεν έχει σημασία πόσα χρήματα ξοδέψαμε στην απασχόληση. Τελικά αυτό που μετράει είναι πόσοι άνθρωποι βρήκαν δουλειά. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να ε, λειτουργήσουμε και να δουλέψουμε πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά. Ας προσπαθήσουμε να αφυπνίσουμε τους νέους, ούτως υπήν. Όσοι εργάζονται στα γραφεία απασχόλησης ε, του εκάστοτε ΟΑΕΔ, ας ε, αναδιπλώσουν, να σηκώσουν τα μανίκια. Ας χαλαρώσουν τις ε, γραβάτες τους, να έρθουν πιο κοντά στους νέους, να καταλάβουν τι χρειάζονται οι νέοι. Οι νέοι μισούν τις ουρές, τις μοναπευθυντικές θηρίδες, τη γραφειοκρατία. Ας καταργήσουμε αυτή τη γραφειοκρατία, ας δώσουμε μια ευκαιρία στους νέους και οι νέοι θα αλλάξουν την Ευρώπη. Ο κύριος Κίτσικη, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Κοιτάξτε, πάρα πολλά ε, Είναι πολύ μεγάλη η ανεργία των νέων σίγουρα και θα πρέπει να έχουμε στοχοθετημένες προσεγγίσεις. Καλωσορίζω αυτή την πρωτοβουλία. Το Φεβρουάριο όμως το 2015 πες σχεδόν 5 εκατομμύρια άνθρωποι νέοι δεν είχαν δουλειά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνω ότι πολλά κράτη-μέλη δυσκολεύονται να ξεκινήσουν τα επιχειρησιακά προγράμματα που αποτελούν την ε, εφαρμογή στην πράξη της πρωτοβουλίας αυτής. Και εγώ ήμουν από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είχαν στηρίξει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αυξήσει την εκ των προτέρων την προκαταρκτική ε, χρηματοδότηση. Ωστόσο αυτό δεν θα λύσει το πρόβλημα από μόνο του. Και γι' αυτό το λόγο ερωτώ το Συμβούλιο τι θα κάνετε επιτέλους για να αποτε... εφαρμοστούν αποτελεσματικά τα μέτρα αυτά και κυρίως πώς θα μετρήσετε τα αποτελέσματα. Πρέπει να σκεφτούμε και να έχουμε υπόψη μας ότι η ανεργία δεν είναι θέμα μόνο έλλειψης θέσεων απασχόλησης. Η ανεργία για πολλούς ε, στην Ευρώπη είναι ένα θέμα διακριτικής μεταχείρισης και ρατσισμού. Οι Ρωμά που αποτελούν ε, το λαό που αντιμετωπίζει τις πιο πολλές ε, διακριτικές μεταχειρήσεις. Ε, τριπλή είναι η ενεργεία μεταξύ των Ρωμά. Ναι, οι Ρωμά ε, έχουν δυσανάλογα μεγαλύτερη ανεργία. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ειδική προσπάθεια για να υποστηρίξουμε τους νέους Ρώμα και θα πρέπει η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων να απευθυνθεί ειδικά και ιδιαίτερα προς τους Ρωμά για να έχουν μια καλύτερη ζωή και να, μπορέσουν, να μπορέσουμε να βάλουμε ένα τέλος σε αυτό το αίσθημα κατά το Ρωμά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι που θέσατε το ερώτημα όσον αφορά την υλοποίηση της πρωτοβουλία στην απασχόληση των νέων. Πολύ σωστά συμπεράνατε ότι χώρες με τη μεγαλύτερη ενεργεία των νέων και οι χώρες εκείνες που επλήγησαν από την κρίση περισσότερο μένουν πίσω όσον αφορά την υλοποίηση ε, της πρωτοβουλίας ανεργία των νέων και την εγγύηση για τους νέους. Η Κροατία είναι σε ύφεση για έξι χρόνια τώρα. Ε, το επίπεδο της ανεργίας των νέων είναι κοντά στο 40%. Σύμφωνα με τα στοιχεία Ευρωστάτ, είναι το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη. Η νεολαία μας φεύγει από την χώρα μας και ψάχνει για δουλειές σε άλλα κράτη-μέρη και η κυβέρνηση δεν χρησιμοποίησε ούτε ένα ευρώ από την πρωτοβουλία μέχρι το Φεβρουάριο του 2015. Η ερώτησή σα ήταν το Συμβούλιο πώς προτίθεται να ενθαρρύνει ταχεία και αποτελεσματική υλοποίηση της πρωτοβουλίας αυτής βραχυπρόθεσμα. Πιστεύω το Συμβούλιο δεν μπορεί να, να προωθήσει τις κυβερνήσεις που είναι ανίκανες να κινηθούν στα κάτι μέλη, μόνο οι ψηφοφόροι να το πετύχουν αυτό. Ευχαριστώ λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε ο κύριο Νέκοφ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Νέκοφ. Ε, κυρία Πρόεδρε, πέρασε ένας χρόνος μετά την εκκίνηση της πρωτοβουλίας, αλλά τα αποτελέσματα στα κράτη-μέλη πόρο απέχουν από τα προσδοκόμενα. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όχι μόνο τα παρόντα οικονομικά εργαλεία που διαθέτουμε, αλλά να προσπαθήσουμε επίσης να κάνουμε μεταρρυθμίσεις όσον αφορά τα συστήματα της παιδείας θα πρέπει να βρούμε νέες μορφές άτυπης ε, κατάρτισης και εκπαίδευσης. Θα πρέπει να βρούμε νέους τρόπους ε, απόκτησης εμπειριών και θα πρέπει να προωθήσουμε ε, καινοτόμο προσέγγιση και προβληματισμό και τρόπο σκέψης στους νέους. Πιστεύω ότι αυτού του είδους η πρωτοβουλία θα πρέπει να προσαρμοστούν δεόντως στα διάφορα κάτι μέλη. Στη Βουλγαρία, παραδείγματο χάρη, μία από τις μεγαλύτερες ε, προκλήσεις είναι η σκληρή μετάβαση από σχολείο προς πανεπιστήμιο. Μαζί με αυτό το πρόβλημα στη χώρα μου πολλοί νέοι μεταναστεύουν. Γι' αυτό πιστεύω ότι το Συμβούλιο δεν θα πρέπει μόνο να προσπαθήσει να βελτιώσει τα προγράμματα αυτά, αλλά θα πρέπει επίσης να, να κινηθεί για ενημέρωση. Ευχαριστώ. Η κυρία Καλίνα Λικασεύσκα έχει το λόγο. Κυρία Προέδρε, αξιότιμα μέλη, δράτω με τις ευκαιρίες να επισημάνω για μία φορά ακόμα Διακόπτεται η ομιλήτρια. Το Συμβούλιο έχει το λόγο, λέει η κυρία Πρόεδρος. Λοιπόν, δράτω με τη ευκαιρία λέγω να επισημάνω εκ νέου τη μεγάλη πολιτική σημασία που έχει η πρωτοβουλία την ενεργεία των νέων. Θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωκοινοβούλιο. Ήταν πολύ καρποφορά συνεργασία μας. Μας επέτρεψε να κινηθούμε τάχιστα, να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της ενεργείας των νέων. Με ρωτήσατε, τι συγκρατεί τα κράτη-μέλη σε αυτή τη φάση. Δύσκολο να αξιολογήσουμε πλήρως την επιτόπια πρόοδο. Και δεν ξεκίνησε ο κύκλος υποβολής εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρα από τα οικονομικά θέματα και τα θέματα οικονομικής ρευστότητας, που είναι πολύ πιεστικά προβλήματα, έχουμε και άλλα προβλήματα. Η ταχεία κινητοποίηση και απορρόφηση των μέτρων. Πρώτα απ' όλα τα κράτη-μέλη δεν έχουν κατάλληλη εφαρμοστική δομή. Δεύτερον, ο καθορισμός των αρμοδίων αρχών. Δημιουργεί προβλήματα σε καποια κάτι κράτη-μέλη. Υπάρχουν και προβλήματα διοικητικού δυναμικού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την υλοποίηση των σχετικών μέτρων της πρωτοβουλίας για τους νέους. Πώς μπορεί να ενθαρρύνει το Συμβούλιο ταχεία εφαρμογή. Το Συμβούλιο πιστεύει όπως και το Ευρωκοινοβούλιο, ότι επαρκής ρευστότητα θα επιτρέψει ταχύτερη εφαρμογή σχετικών μέτρων πολιτικής που καθορίζονται στα εθνικά σχέδια. Η νέα πρόταση για την αύξηση προχρηματοδότησης θα πρέπει να συμβάλλει σε ταχύτερη κινητοποίηση των πόρων. Έτσι, θα αυξηθεί η δυνατότητα των εθνικών αρχών να ξεκινήσουν διαγωνισμούς για προγράμματα και να επεξεργάζονται τις αιτήσει ταχύτερα. Η πρόσθετη συγχρηματοδότηση θα καταβάλλεται στα κρατη μέλη αμέσως μετά τη θέση ισχύ του τροποποιητικού κανονισμού. Θετικός αντίκτυπος πρέπει να αναμένεται σύντομα. Η εφαρμογή του, ε, της εγγύσης του νέους χρειάζεται και διαθοντικές μεταρρυθμίσεις και μέτρα που εφαρμόζονται τομικό επίπεδο. Τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν κράμα εθνικών πολιτικών για την ενεργεία των νέων βάσει των συγκεκριμένων αναγκών τους και προτεραιοτήτων τους. Η εγγύηση για τους νέους είναι ένα από τα μέτρα. Όλα τα κράτη-μέλη υπέβαλαν τα εφαρμοστικά του σχέδια για την εγγύηση των νέων και εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο παρακολουθείται τεχνικά από το Συμβούλιο. Βασιζόμαστε σε, στη συμβολή της Επιτροπής Απασχόλησης. Κινούμεθα πολυμερώς, με βάση δείκτες και τις ειδικές διαδικασίες. Ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ κρατών μελών και αυτή είναι σημαντική. Και αξιολόγηση αποτελεσμάτων των μέτρων που εφαρμόζονται. Κλείνοντας, να υπογραμμίσω κάτι. Τα κράτη-μέλη υποβάλλουν δομημένα στοιχεία στις εκθέσεις τους για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας στην ανεργία των νέων. Οι εκθέσεις θα δώσουν μια σφαιρική εικόνα της σας πρόοδου των κρατών μέλων για την εφαρμογή των πρωτοβουλίων αυτών. Έτσι θα τροφοδοτηθεί η ανάλυση του Συμβουλίου για περαιτέρω μέτρα που χρειάζονται και θα γίνεται και ο τακτικός έλεγχος Συμβουλίου. Ο αποτελεσματικός έλεγχος είναι προϋπόθεση επιτυχούς εφαρμογής και συνέχεια της ορθής χρηματοδοτήσεω. Σε σχέση με αυτό, το Συμβούλιο, εδραζόμενο επί του έργου της Επιτροπής Απασχόλησης, ακολουθεί πολυμερή επιτήρηση της εφαρμογής και γίνεται ανάλυση ομοτήμων των μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιούνται και που συμπεριλαμβάνονται στις συστάσεις κατά χώρα. Τέλος, βάσει των εμπειριών του 2014 και με μικρή βελτίωση των στοιχείων ενεργεία των νέων στα κράτη-μέλη που πλήττονται σκληρότερα, πρέπει να αναμένεται ότι το ζήτημα αυτό θα εξεταστεί στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2015. Εν πάση περιπτώσει, το Συμβούλιο θα συζητήσει ενδελεχέστερα το θέμα στη Σύνοδο του Ιουνίου μαζί με την ειδική ε, έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν περαιτέρω και τις προσπάθειες που καταβάλουν και θα πρέπει να κάνουν διαθετικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται και να εφαρμόσουν ποιοτικά μέτρα για να συμμετάσχουν οι νέοι έτσι στις αγορές εργασίας μέσω εκπαιδεύσεως και αυτά είναι σημαντικότατα μέτρα. Συνοψίζοντα. το Συμβούλιο και αυτό συμφωνεί ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα. Περισσότερα για να καταπολεμηθεί η ανεργία των νέων. Παρέθεσα κάποια παραδείγματα μέτρων που έχουν δρομολογηθεί στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχουν σαν στόχο το σύστημα να γίνει αποτελεσματικότερο. Δεν μπορώ να σα υποσχεθώ θαύματα και ότι θα γίνει το θαύμα αύριο, αλλά μπορώ να πω ότι έγινε σκληρή δουλειά. Προσπαθήσαμε να βρούμε λύση το ταχύτερο δυνατόν. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία μου. Πέρα